I uh, Να αρχίσουμε παρακαλώ. Έχω τόσο πολλά να διαβάσω εδώ ως ανακοινώσει. Ε, καλώς ήρθατε στη συνεδρίαση. Η διερμηνία είναι σε δύο... Ε, η συνεδρίαση είναι σε δύο τμήματα. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10.30 και θα έχουμε τις συστάσεις για απόφαση του Συμβουλίου για να ε, ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για μια Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την πρόληψη της τρομοκρατίας με βάση το άρθρο 218 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ξένους μαχητές όπως το αποκαλούμε μετά το επόμενο τμήμα της συνεδρίασης της ΛΥΜΠΕ θα είναι κοινή συνεδρίαση με την ΤΕΒΕ στις 10.40 στην αίθουσα Αλτιέρος Σπινέλη 3G3. Τώρα, για αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη, το Συμβούλιο της Ευρώπης προετοιμάζει ένα συμπληρωματικό πρωτόκολλο στη Σύμβαση για την Πρόληψη Τρομοκρατίας για να εφαρμόσει το ψήφισμα 278 για του τρομοκράτε ξένου μαχητέ που εγκρίθηκε τον προηγούμενο Σεπτέμβριο από το Συμβούλιο Ασφαλεία των Ηνωμένων Εθνών. Το πρωτόκολλο αυτό το οποίο συμφωνήθηκε σε μια σύντομη περίοδο θα καταστήσει ποινικό αδίκημα την ε, ε, ε, εκπαίδευση για τρομοκρατία, την οργάνωση, τη χρηματοδότηση και το ταξίδι για τρομοκρατία με βάση το άρθρο 218 τη συνθήκη. για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τις εσωτερικές αρμοδιότητε τη Ένωση λόγω του ότι υπάρχει απόφαση, για το πλαίσιο, απόφαση πλαίσιο για τρομοκρατία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε συστάσει για μια απόφαση του Συμβουλίου για να εγκριθεί η έναξη διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με το άρθρο 218, το Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει τη σύμφωνη γνώμη του για να συμφωνηθεί το πρωτόκολλο αυτό και λόγω τη επιπτώσεις που θα είχε για την απόφαση πλαίσιο για την δημοκρατία. Γι' αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό το Κοινοβούλιο να συμμετάσχει σε αυτέ τις διαπραγματεύσει. Γι' αυτό έχουμε εδώ σήμερα μαζί μας ε, την Επιτροπή που θα παρουσιάσει τη συστάση τη για μια απόφαση του Συμβουλίου για εντολή διαπραγματεύσεων και καλωσορίζουμε τον κύριο Κουέτζικοφ, ο οποίο είναι ο συντονιστής ε, κατά τη τρομοκρατία του Συμβουλίου τη Ευρώπη που θα παρουσιάσει το πλαίσιο και το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων. Οπότε πρώτα να δώσω το λόγο στον κύριο Ολιβιέ Λουίκ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ που μας καλέσατε εδώ σήμερα το πρωί για να σας ενημερώσουμε για το πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Όπως και εσείς ήδη είπατε, η προσπάθεια η οποία ξεκίνησε στο Συμβούλιο της Ευρώπης από τον προηγούμενο Ιανουάριο προέρχεται, βασίζεται από την απόφαση Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις 24 Δεκεμβρίου. Έγινε μια συνεδρίαση στις 17 Σεπτεμβρίου του Συμβουλίου Ασφαλείας σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στη Νέα Υόρκη. Το ψήφισμα λοιπόν του Συμβουλίου Ασφαλείας υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να ποινικοποιήσουν ορισμένες συμπεριφορές και ορισμένα είδη επαφών πολιτικών που συνδέονται με το φαινόμενο των ξένων μαχητών, αλλοδαπών μαχητών. Εμείς εξετάζουμε το θέμα αυτό σε επίπεδο επιτροπής εδώ και αρκετό καιρό και το θέμα το οποίο έχει ήδη συζητηθεί αλλά και στο Συμβούλιο είναι το εάν θα πρέπει να διευρύνουμε και να λισαβονοποιήσουμε σε εισαγωγικά τις ρυθμίσεις για την καταπολέμηση των ξένων μαχητών. Αυτό ξεκίνησε το 2002 και ολοκληρώθηκε το 2008. Ε, τα πράγματα εξελίχθηκαν με τέτοιο τρόπο όμως που το, η Υπουργική Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης την 21η Ιανουαρίου σε ένα πλαίσιο οξυ, αντίληψης οξυμένων επιθέσεων, θυμάστε τι είχε γίνει στη Γαλλία κτλ, αποφάσισαν να προχωρήσουν με υψηλότερη ταχύτητα. Θεωρούμε σε επίπεδο διαδικασίας ότι βρισκόμαστε σε μια κάπως περίεργη κατάσταση, γιατί έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων στο Στρασβούργο, και εμείς εξακολουθούμε να συζητάμε κατά της εντολής την οποία δίδουμε. Στην ουσία δηλαδή στοχεύουμε σε ένα κινούμενο στόχο. Οι εκπρόσωποι που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις στο Στρασβούργο προσπαθούν να συντονίσουν κατά κάποιο τρόπο τις θέσεις των κρατών μέλων με τις θέσεις των υπολείπων εμπλεκομένων. Και γι' αυτό δημοσιεύσαμε και μία πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τις κατευθυντήριες γραμμές. Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι συνοπτικές, σύντομες, βασίζονται στο άρθρο 218 στο 2.18 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκινάμε από την αξιολόγηση η οποία γίνεται ότι αν όχι το σύνολο, τουλάχιστον ένα μεγάλο τμήμα των θεμάτων τα οποία συζητάμε στα πλαίσια της πρότασης του κοινού πρωτοκόλου, είναι αρμοδιότητα κοινοτική, ενωσιακή μάλλον. στόχος είναι να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περαιτέρω ποινικοποίηση ορισμένων συμπεριφορών εφόσον αυτές οι συμπεριφορές εξελίσσονται, θα έλεγα εφαρμόζονται με στόχο την στράτευση, την προετοιμασία, την παθητική εκπαίδευση για τρομοκρατικές ενέργειες. Ε, τα ταξίδια ή την προσπάθεια ταξιδιού και μετακινήσεων για λόγους τρομοκρατικούς, ε, προσπάθειες επηρεασμού ε, φύλων και στην ουσία αυτό είναι το τι διαπραγματευόμεθα. Το νομικό τμήμα είναι σύντομο, είναι τρεις παράγραφοι. Λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαπραγματευτεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη-μέλη θα πάρουν μέρος στις διαπραγματεύσεις και θα υπάρξει συντονισμός στην Επιτροπή ad hoc, δηλαδή στο Συμβούλιο στην Αρμόδια Επιτροπή. Όπως επίσης θα υπάρξει και ad hoc συντονισμός. Κάναμε και τα δύο. Πρέπει να ευχαριστήσω την Προεδρία, να ευχαριστήσω τα κράτη-μέλη για την ευελιξία τους στην αντιμετώπιση του θέματος αυτού με σύντομο τρόπο. Και υπήρξε ad hoc συντονισμό στο Στρασβούργο πριν από τις συναντήσεις της διαπραγματευτικής ομάδας. Οι προπαρασκευαστικές αυτές συναντήσεις πήγαν καλά και υπάρχει μια σαφής θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα οι οδηγίες, οι διαπραγματευτικές οδηγίες υπενθυμίζουν ότι το θέμα είναι η εφαρμογή υποχρεώσεων που προέρχονται από το κεφάλαιο 7 της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών. Το κομβικό θέμα, η ουσία αν θέλετε, είναι η ποινικοποίηση των συμπεριφορών, τις οποίες μόλις υπενθύμησα συμπεριφορές οι οποίες διαπιστούνται στην λειτουργική παράγραφο υπαριθμός 6 του Συμβουλίου, της, ε, της απόφασης του Συμβουλίου, του ψηφίσματος μάλλον του Συμβουλίου. Και επίσης ε, ε, μπορεί να χρησιμοποιηθούν αν χρειαστεί και άλλα τμήματα του συγκεκριμένου ψηφίσματος εφόσον είναι απαραίτητο για να αντιμετωπιστούν τα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην παράγραφο 6. Υπάρχει λοιπόν μια σαφής εντολή. Εφόσον αυτό χρειαστεί βέβαια, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τις παραγράφους 4 και 5. Οι κατευθυντήριες γραμμές τις οποίες ακολουθούμε και τις οποίες προτείνουμε στη συγκεκριμένη αυτή οδηγία είναι πρώτον ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στην σύμβαση αυτή θα πρέπει να ποινικοποιήσουν τις συγκεκριμένες ε, ε, συμπεριφορές στο εθνικό τους επίπεδο σεβόμενοι πλήρως το κοινοτικό και εκτιμένο. Δεύτερον, νομική βεβαιότητα και προβλεψιμότητα πρέπει να διασφαλιστεί και κανένα εμπλεκόμενο μέρος, κανένα κράτος μέλος δεν θα πρέπει να ποινικοποιήσει και να δημιουργήσει νέου τύπου ποινικέ συμπεριφορές εφόσον στο εσωτερικό σύστημα νομικό υπάρχουν αντίστοιχες προβλέψεις. Δεν χρειάζεται δηλαδή να υπάρχουν επικαλύψεις. Συνεπώς λοιπόν έχουμε κάποιο περιθώριο για την προσπάθεια που θα πρέπει να γίνει σε εθνικό επίπεδο και σε ενωσιακό επίπεδο. Μπορούμε να αποφασίσουμε, μπορούμε να κρίνουμε ε, αν θα πρέπει κάποιες ενέργειες, κάποιες πράξεις να ποινικοποιηθούν εκ νέου ή σε εθνικό επίπεδο έχουμε ήδη τα μέσα τα οποία απαιτούνται για την αντιμετώπιση τους. Και τέλος, υπάρχει και η ρήτρα ανάδρασης που περιλαμβάνονται στο άρθρο 26 της αρχικής σύμβασης, της μητρικής σύμβασης του 2005 που ετέθησε λειτουργία το 2007. Λέγεται εκεί ότι στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυρίαρχο νομικό επίπεδο είναι ο κοινοτικό νόμος, η κοινοτική νομική τάξη. Λοιπόν, αυτά για την εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Σας... Ευχαριστούμε πολύ. Ε, Πρώτα θα δώσω το λόγο στην, την Πρόεδρο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ και καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που μου δώσατε το λόγο και ευχαριστώ που με προσκαλέσατε. Πράγματι θέλω να σας ενημερώσω για την κατάσταση πραγμάτων όσον αφορά την εντολή στο Συμβούλιο. Η Προεδρία γνωρίζει ότι οι χώρες μέλη έχουν κατανοήσει πολύ καλά την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Όπως είπε και ο το Συμβούλιο της Ευρώπης λοιπόν άρχισε να εργάζεται πάνω σε ένα πρωτόκολλο αρκετά γρήγορα και προχώρησε αρκετά γρήγορα, είναι αλήθεια. Από την πλευρά μας περιμέναμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρθει με εντολή και μόλις πήραμε την εντολή, η Προεδρία θεώρησε ότι είναι ιδιαίτερα επίγον ζήτημα και προχωρήσαμε έτσι πάρα πολύ γρήγορα. Είχαμε δύο συμβούλια Υπουργών Δικαιοσύνη προκειμένου να καταλήξουμε στην εντολή και να είναι εντολή αποδεκτή από όλου. Συζητήσαμε περισσότερο την εντολή παρά τις κατευθυντήριες γραμμές στην αρχή και υπήρξαν κάποια θέματα σημαντικά και για τις χώρες μέλη. Συνεχίσαμε λοιπόν με τον ίδιο τρόπο όπως ε, είχαμε κάνει τη συζήτηση και στο Συμβούλιο της Ευρώπης με τη συμμετοχή των χωρών μελών, με διαπραγματεύσεις και θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Οι χώρες μέλη κατάλαβαν επίσης ότι δεν θέλουμε να παρατείνουμε τη συζήτηση στο Συμβούλιο της Ευρώπης, γι' αυτό και προχώρησαν γρήγορα σχεδιάζουν και εδώ ο συνάδελφός μου εκ δεξιών θα το επιβεβαιώσει ποια είναι η κατάσταση στο Συμβούλιο. Πάντως ήδη τον Μάιο σκοπεύει το Συμβούλιο της Ευρώπης να τον κρίνει. Οι χώρες μέλη κατάλαβαν ότι η εντολή αυτή χρειάζεται γρήγορα. Γενικά μιλώντας λοιπόν η Προεδρία κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να οριστικοποιηθεί η εντολή και ελπίζουμε να έχουμε σήμερα κάποια απόφαση και στην επόμενη συνεδρίαση στο Συμβούλιο της Ευρώπης που θα γίνει στις 7 Απριλίου, μετά το Πάσχα δηλαδή, θα έχουμε, πιστεύουμε, εντολή τη, για συμμετοχή της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διαπραγματεύσεις. τους κβό λοιπόν από πλευράς της Προεδρίας. Και η προσέγγιση μας είναι ιδιαίτερα θετική και για την Προεδρία και για τις χώρες μέλη. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο με τον ίδιο τρόπο όπως το έχουμε κάνει και κατά το παρελθόν. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Τώρα ο κύριος Κουέτζικοφ έχει το λόγο που είναι ο συντονιστής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας να μας μιλήσει για το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα. Η συζήτηση για την τρομοκρατία στην Επιτροπή σα δεν γίνεται υπό την απειλή κάποιας τρομοκρατίας. Βέβαια δεν είναι ότι θα τον αναγνωρίζετε μπαίνοντα μέσα ο τρομοκράτη αμέσω, θα βλέπατε ότι είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε ασφαλεί κατά τη διάρκεια τη συζήτηση αυτή εδώ. Θέλω λοιπόν να μιλήσω στην ΛΥΜΠΕ Λίμπε την ξέρουμε όλοι. Δεν ξέρουμε τι ακριβώ σημαίνει το Λίμπε, αλλά ω Λίμπε την ξέρουμε. Εν πάση περιπτώσει, είμαι ευγνώμων στην Επιτροπή και στην Προεδρία για την ε, μεγάλη πολιτική στήριξη. Το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια όλων των διαπραγματεύσεων του πρόσθετου πρωτοκόλου βρεθήκαμε σε κάπως έκτακτη κατάσταση. Αντιδρούμε στο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, πρόκειται για το κεφάλαιο 7, του χάρτη όσον αφορά την τρομοκρατία. Είναι το δεύτερο ψήφισμα. Το πρώτο εγκρίθηκε λίγο μετά την 10η Σεπτεμβρίου ως αντίδραση στην τρομοκρατική επίθεση που έγινε τότε στη Νέα Υόρκη. Αυτό είναι το δεύτερο τέτοιο ψήφισμα λοιπόν. Πριν περάσω στο πρωτόκολλο αυτό καθε αυτό, θα ήθελα να αναφέρω δύο-τρία λόγια για το τι κάνει για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Οι διάφορες οργανώσεις το βλέπουν διαφορετικά θέμα εθνικής ασφάλειας για τα Ηνωμένα Έθνη. Για μας είναι απειλή στη, στα δημοκρατικά καθεστώτα των χωρών μελών μας. Ξεκινήσαμε από το 1978, όταν οι δηλώσεις ήταν μια σελίδας όλες και όλες. Και τότε είπαμε ότι η τρομοκρατία είναι απειλή στη δημοκρατική τάξη των χωρών μελών μας. Μετά είχαμε τη διάσκεψη της Βαρσοβίας το 2005 που και εκεί εγκρίθηκε μία πρόταση που ισχύει πάντα που λέει ότι η τρομοκρατία είναι απαράδεκτη κατά οποιασδήποτε συνθήκες και σε οποιοδήποτε πολιτιστικό πλαίσιο. Έτσι λοιπόν η προσέγγιση μας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας είναι ότι πλήττει τη δημοκρατία και ότι είναι απαράδεκτη. Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών εγκρίναμε διάφορες συμβάσεις. Έχουμε και παλιότερες για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Έχουμε το θέμα της πρόληψης και του χειρισμού που είναι πολιτικό αδίκημα και οδηγεί σε έκδοση του τρομοκράτη, αυτά στη δεκαετία του 70. Στη συνέχεια έχουμε και την αρχική σύμβαση του πρωτοκόλου που είναι η Σύμβαση για την Πρόληψη της Τρομοκρατίας, η οποία όταν εγκρίθηκε ήταν μια καινοτομία, διότι ζητούσε από τα κράτη-μέλη να ποινικοποιήσουν την προετοιμασία κάποιων τέτοιων ε, αδικημάτων τρομοκρατίας. Είτε πρόκειται για την, ε, την ενθάρρυνση, για τρομοκρατικές πράξεις ε, κτλ. Έχουμε επίσης για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την χρήση ειδικών ερευνητικών πρακτικών στις ανακρίσεις σοβαρών αδικημάτων και τρομοκρατίας. Το Συμβούλιο της Ευρώπης βέβαια στηρίζει απόλυτα τα ανθρώπινα δικαιώματα για όλους. Για τα θύματα, και για τους τρομοκράτες. Θα θυμόσαστε ότι οι συνάδελφοί σας από το Συμβούλιο της Ευρώπης όταν υπήρξε εκείνο το πρόγραμμα της CIA για τις ε, παράνομες μεταφορές κρατουμένων θα θυμόσαστε ότι στηρίξαμε την έννοια ότι πρέπει να τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα και όταν καταπολεμούμε την τρομοκρατία. Θυμάμαι και τους δικούς σας υπουργούς και πρέσβεις που είπαν ότι όχι δεν κάνουμε τέτοια μέχρι που ο πρόεδρος Μπούς είπε ναι υπήρξε τέτοιο πρόγραμμα. Συνεπώς εμείς και το δικαστήριό μας θα στηρίξει πάντα τα ανθρώπινα δικαιώματα οποιοδήποτε ισχυρίζεται ότι ήταν θύμα τέτοιας παραβίασης. Αυτό είναι επίσης κάτι πολύ σημαντικό για μας, η υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε και μια άλλη σημαντική γραμμή και αυτή είναι η αμοιβαία συνδρομή. Έχουμε 20 περίπου τέτοιες συμβάσεις. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα. Εμείς δεν έχουμε το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης κλπ. Αλλά όταν πρόκειται για την τρομοκρατία, δεν αφορά μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση, πάμε και πιο μακριά. Και έτσι ερχόμαστε και στους ξένους μαχητές. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε στη διάθεσή μας αυτόν τον εξοπλισμό. Και τέλος, Ό,τι κάνει το Συμβούλιο της Ευρώπης για να ενθαρρύνει τον διαπολιτιστικό διάλογο, τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, όλα αυτά μπορούν να προλάβουν τις συνθήκες εκείνες οι οποίες οδηγούν στην τρομοκρατία. Τώρα έρχομαι στο πρωτόκολλο αυτό καθε αυτό ανέφερα ότι υπάρχει πολιτική αναγκαιότητα για αυτό το πρωτόκολλο και χαιρόμαι πολύ που είχαμε τόσο ευρεία ε, πολιτική στήριξη. Πρέπει επίσης να σας πω εδώ ότι το πρωτόκολλο το διαπραγματευτήκαμε με απόλυτη διαφάνεια. Μέχρι τώρα η δική ομάδα εργασίας που έκανε τις διαπραγματεύσεις συνεδρίασε τρεις φορές. Μετά την πρώτη συνεδρίαση αποφάσισαν ότι κάθε σχέδιο που είχαν, θα το δημοσιοποιούσαν. Μόνο δεν δημοσιοποιήθηκε εκείνο το κείμενο το οποίο από κάτω είχε κάποιες ε, υποσημειώσεις για ειδικέ θέσεις των κρατών μελών. Όταν αυτές απαλήφθηκαν δημοσιοποιήθηκε και αυτό το κείμενο. Ενημερώθηκαν και η Διεθνής Αμνηστία και η Διεθνής Οργάνωση Νομικών είχε πρόσβαση στο πρωτόκολλο αυτό και έχουμε μια διαδικασία όπου αν το ζητήσουν μπορούν να έρθουν παρατηρητές στις εργασίες της ομάδας αυτής της εργασίας. Δεν χρησιμοποίησαν αυτή την ευκαιρία. Η Επιτροπή μας όμως αυτό που έκανε ήταν ότι δημοσιοποίησε το πρωτόκολλο και σε εκείνους. Με αποτέλεσμα να πάρουμε διάφορα σχόλια από αυτούς, τα οποία και χρησιμοποίησαμε και συμπεριλάβαμε. Επί της ουσίας τώρα. νομικά είναι ένα πολύ λεπτό και το θέμα. Γιατί κάθε αδίκημα ε, σημαίνει ότι υπάρχει μια πράξη και υπάρχει και μια πρόθεση. Και σύμφωνα με τα δικά μας νομικά καθεστώτα δεν είναι η πρόθεση που αποτελεί αδίκημα αλλά η πράξη. Όταν λοιπόν προετοιμάζεται μια τρομοκρατική πράξη, η πρόθεση έχει μεγάλη σημασία και γι' αυτό θέλουμε να πλησιάσουμε όσο γίνεται περισσότερο την πρόθεση. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε πάντα με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένα από τα θέματα που αντιμετωπίζουμε, που αντιμετωπίσαμε μάλλον, βγήκε από το πρωτόκολλο, δηλαδή η προσπάθεια να ποινικοποιήσουμε το γεγονός ότι κάποιος προσλαμβάνεται για να κάνει μια τρομοκρατική πράξη. Δεν υπάρχει πια στο πρωτόκολλο γιατί σε τρεις ε, συνεδριάσεις η ομάδα εργασίας δεν βρήκε τη νομική βάση για να το συμπεριλάβει. Ίσως αν είχαν γίνει 10-20 συνεδριάσει να είχαν βρει μια λύση. Προ το παρόν πάντως δεν συμπεριλαμβάνεται. Όπω είπε και ο συνάδελφο, κάποιες χώρες μέλη πήγαν πιο μακριά από το πρωτόκολλο. Για το άρθρο 2, για παράδειγμα, το οποίο λέει στην περίπτωση που κάποιος ε, γίνει μέλος σε μια οργάνωση που σκοπεύει να προβεί σε κάποια δίκημα. Πρόκειται για θέματα συνομασίας, ασοσιασιών de malfaiteur. Κάποιες από τι χώρε μέλη λοιπόν πήγαν πιο πέρα. Η Γαλλία για παράδειγμα η ΣΥΓΑΓΕ, το Entreprise να de δηλαδή μια ιδιωτική ατομική επιχείρηση για τρομοκρατία. Το πρωτόκολλο δεν φτάνει στα άκρα, αν μπορώ να το πω έτσι, ενώ άλλες χώρες μέλη το έκαναν. Πάντω η προστιθέμενη αξία του πρωτοκόλου μεταξύ άλλων είναι και το ότι εναρμονίζει όσο γίνεται περισσότερο την υπάρχουσα νομοθεσία. Όταν φτάνουμε στα θέματα έκδοση, υπάρχει το θέμα της διπλής εγκληματικότητα, Αν ένα αδίκημα δεν είναι στην χώρα από την οποία ζητιέται, δεν μπορεί να υπάρξει έκδοση. Προσπαθούμε να αποφύγουμε λοιπόν τη διάδοση της τρομοκρατίας και τους ξένους μαχητές. Είπαμε ότι ποινικοποιείται η κατάρτιση για τις τρομοκρατικές πράξεις, η διευκόλυνση τέτοιων ξένων μαχητών εφόσον σκοπεύουν να προβούν σε κάποια τρομοκρατική πράξη και υπάρχει και το άρθρο 7 που μιλάει για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών. Είναι μια μεγάλη προστιθέμενη αξία, πιστεύω, στο πρωτόκολλο. Γιατί τα συμβαλόμενα μέρα, μέρη πρέπει να ορίσουν συγκεκριμένα σημεία επαφής για την ανταλλαγή πληροφοριών. Στην πράξη δηλαδή, αν μια χώρα, για να τα πω τα πράγματα με το όνομα του, αν η Τουρκία σταματήσει κάποιο στα σύνορα γιατί υποπτεύεται ότι αυτός πάει στη Συρία, τότε πρέπει να μπορεί, αν είναι αυτός πολίτης Ευρωπαϊκής Ένωσης, να καλέσει κάποιον και να πάρει πληροφορίες. Να ελέγξει στο μεταξύ το διαβατήριο, τελωνία, ελέγχου κτλ. Και στο μεταξύ παίρνει αυτή την πληροφορία. Γιατί αν δεν πάρει αυτή την πληροφορία, είναι υποχρεωμένη η Τουρκία να αφήσει το άτομο αυτό να συνεχίσει προ ε, τον προορισμό του. Αυτή λοιπόν η ταχεία ενημέρωση πρακτικά γίνεται δυνατή. Μην πω τώρα στις νομικές λεπτομέρειες για τους ορισμούς. Σας διαβεβαιώ ότι περισσότερες συζητήσεις που έγιναν στις διαπραγματεύσεις επικεντρώθηκαν ακριβώς σε αυτό. Πώς δηλαδή να προστατεύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, ποινικοποιώντα όμως αδικήματα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε τρομοκρατικές επιθέσεις. Κυρίως όσον αφορά τους ξένους μαχητές. Πράγματι στο πρωτόκολλο το άρθρο της Αρχικής Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συμπεριλήφθηκε εδώ. Έτσι αποφάσισαν οι συντάκτες του κειμένου. Οι φίλοι μας από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις θέλησαν οι συντάκτες να συμπεριλάβουν περισσότερα πράγματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι συντάκτες όμως αποφάσισαν ότι αν αρχίσουμε να διευρύνουμε τον κατάλογο, τότε μπαίνουμε στο ζήτημα της ερμηνείας του γιατί κάτι το οποίο ισχύει δεν υπάρχει μέσα. Οπότε συμπεριέλαβαν τα πιο σημαντικά. Τα υπόλοιπα εννοούνται. Έτσι τουλάχιστον ήταν το πνεύμα των συντακτών. Όσον αφορά τη διαδικασία, στο Συμβούλιο της Ευρώπης το πρωτόκολλο έχει προχωρήσει, δηλαδή έχει συνταχθεί μετά τις τρεις αυτές ε, συναντήσεις και τώρα το πρωτόκολλο πάει στην Επιτροπή Ειδικών επί της Τρομοκρατίας. Υπάρχουν και στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Είναι η Επιτροπή Κολεξτέρ. Είναι οι εμπειρογνώμονες για την τρομοκρατία. Είναι μια επιτροπή, steering committee, η οποία θα εξετάσει το πρωτόκολλο αυτό την εβδομάδα 7 Απριλίου. Και στη συνέχεια θα πάει στην ομάδα εργασίας των ε, Υπουργών ε, Νομικών Υποθέσεων. Είναι εκεί η αρμόδη πρέσβης των ε, νομικών υποθέσεων και στη συνέχεια θα έχουμε τη γνωμοδότηση της Νομικής Επιτροπής, της δικιάς μας Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης. Ο εισηγητής έχει ήδη οριστεί και τέλος θα πάει στην Επιτροπή των Υπουργών προς έγκριση. Η έγκριση θα λάβει χώρα στις 29 Απριλίου κατά πάσα πιθανότητα. Και στις 19 Μαΐου που έχουμε υπουργική ε, συνέλευση εδώ στις Βρυξέλλες, ελπίζουμε ότι κάποιες χώρες τουλάχιστον θα υπογράψουν και μετά θα υπάρξει και η εκδήλωση για την υπογραφή. Τρεις εβδομάδες πριν την έγκριση και την ε, εκδήλωση αυτή, Πρέπει να ξέρετε ότι έτσι καλλιώς οι υπουργοί πρέπει να περάσουν από κάποιες διαβουλεύσεις ορισμένοι τουλάχιστον να μιλήσουν με άλλους υπουργού μερικέ φορέ με τα κοινοβούλια τους. Το χρονοδιάγραμμα είναι αυτό λίγο πολύ. Και πάλι, πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε γρήγορα να εγκριθεί δηλαδή γρήγορα το πρωτόκολλο. Βέβαια το πρωτόκολλο δεν πρόκειται να κάνει καμιά επανάσταση σε σχέση με αυτά που ήδη έχουν εγκριθεί κυρίως από κάποιες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μάλιστα μερικές πάνε και ακόμα πιο μακριά. Πάντως η προστιθέμενη αξία του είναι ότι διευκολύνει τη συνεργασία μέσω αναρμόνισης της νομοθεσίας και πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ σημαντικό αυτό γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, οι χώρες που γετνιάζουν με την Συρία παίζουν σημαντικό ρόλο, πρέπει να παίξουν σημαντικό ρόλο. Και υπάρχει και αυτό το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών που ονομάζεται 24-7. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Κουέτζικοφ. Πολλοί συνάδελφοι θέλουν να παρέμβουν. Να, να πω ποιοι είναι. Mrs. Ravo Dallon, Mr. Uh, Lopez Aguiar, uh, Mrs. Sargentini, Mrs. Gomez, Mrs. Meyer, uh, Mrs. Fayon. If nobody else... Αν δεν υπάρχει άλλος, τότε να κλείσω τον κατάλογο και να δώσω το λόγο. Α, και άλλοι. Α, όχι, όχι, όχι, εντάξει. Α, μόλις μου είπαν ότι πρέπει να σας παρακαλέσω να τηρήσετε χρόνο δύο λεπτών αλλά θα είμαι γενναιόδορη. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε να τελειώσουμε 10 και 30, γιατί 10 και 40 πρέπει να αρχίσει η άλλη συνεδρίαση με συμμετοχή μας. Οπότε, συνάδελφοι, η κυρία Ιντφέλτ. Ευχαριστώ. Ανησυχώ λιγάκι από αυτά που ακούω. Γιατί έμεσα ο κύριος Κούτζικοφ ανέφερε μερικές από τις ανησυχίες μου για τη διαδικασία. Και εσείς εκφράσατε ανησυχίες για τη χρονική αλληλουχία. Η Επιτροπή περιέγραψε με πολύ ασάφεια, τρομερή ασάφεια την διαπραγματική εντολή. Είναι σαν να λέγει υπογράψτε και μετά θα γράψουμε από πάνω τι έχει. Εγώ νομίζω ότι η ουσία αυτής της συμφωνίας επίσης προκαλεί ανησυχίες. Όλοι συμφωνούμε με το στόχο. Όλοι ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Αλλά παρόλα αυτά έχω την εντύπωση ότι κινδυνεύουμε να πάμε προς λάθος κατεύθυνση. προτείνουμε ένα νομοθέτημα το οποίο στοχεύει μόνο ένα τμήμα των τρομοκρατών. Άρα θα έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και συμφωνώ και με αυτό που είπε ο κύριος Κούτζικοφ. ποινικοποιούμε μια πρόθεση. Άμα το διαβάσετε προσεκτικά, ποινικοποιούμε κάποιες ενέργειες, αλλά το να ταξιδέψει κανείς να πάει κάπου με την πρόθεση να εκπαιδευτεί ή να διαπράξει, ε, τι πάει να πει τώρα αυτό, πώς αποδεικνύεται και να πας πού δηλαδή. Άμα πας από τη Βόνη, για παράδειγμα, ξέρω εγώ πού να πας, ε, στο Βερολίνο, για να κάνεις κάποια εγκληματική ενέργεια τι είναι αυτό το ότι πας από τη Βόνη στο Βερολίνο είναι ε, ποινικό αδίκημα και αυτή η έννοια ξένοι μαχητές ε, δεν την καταλαβαίνω αλλά τι πάνε να πει ξένοι μαχητές είναι πολίτες της Ένωσης συμφωνώ με την ανταλλαγή πληροφοριών πολύ σημαντικό τμήμα Καταλαβαίνω γιατί η χρηματοδότηση ή η οργανωτική στήριξη είναι ενέργειες. Καταλαβαίνω ότι αυτά μπορούν να ποινικοποιηθούν. Αλλά ανισχώ ιδιαίτερα για την ποινικοποίηση προθέσεων. Αν κάποιος λοιπόν πάει στο Πακιστάν με τη σαφή πρόθεση να γίνει τρομοκράτης αλλά μόλις φτάσει εκεί σκέφτεται όχι δεν θέλω και επιστρέφω Εν τω μεταξύ τον έχουμε, έχουμε ποινικοποιήσει την πρόθεσή του. Ενώ θα μπορούσε να επανέλθει και να μην γίνει τελικά τρομοκράτης. Χάνουμε αυτή τη δυνατότητα. Θα ήθελα να μας πει η Κομισιόν ε, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, ποια θα είναι η διαδικασία και πώς θα αντιμετωπίσετε τις ανησυχίες μου για την ποινικοποίηση προθέσεων. Ευχαριστώ κύριε Αντιφελείο Πρόεδρος. Θέλω να ενημερώσω ότι δεν έχουμε σήμερα διερμηνία από ή προ τα εστονικά. Για τον κυρία Λόριστο μόλις μπήκε. Η κυρία Βέμβα. Ευχαριστώ πολύ. Στις 24 Σεπτεμβρίου παρελθόντος έτους, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε ένα ψήφισμα για συγκρούσεις και ξένους μαχητές και την τρομοκρατία. Και έκτοτε έχει υπάρξει ένα συμπληρωματικό πρωτόκολλο που μπορούμε να αξιοποιήσουμε στα πλαίσια της διεθνούς συνεργασίας κατά αυτών των εγκλημάτων. Η εργασία αυτή βασίζεται στο άρθρο 83 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το έγγραφο επιτρέπει περαιτέρω διαπραγματεύσεις και μέτρα για την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας. Είναι λοιπόν βήμα, πιστεύω, προ τη σωστή κατεύθυνση το ψήφισμα δεν καθορίζει επακριβώς ποια είναι τα χαρακτηριστικά της τρομοκρατίας αναφέρεται σε ορισμένα είδη συμπεριφοράς, ταξίδια σε άλλες χώρες και κατάρτιση για τρομοκρατία, συμμετοχή σε συγκρούσεις, αλλά δεν υπάρχει ένας ε, συνολικός ορισμός που να μας επιτρέψει να ε, έχουμε ένα κείμενο που να έχει νομικές συνέπειες. Χρειαζόμαστε νομική ασφάλεια στην κοινωνία μας. Πρέπει να ξέρουμε ποιες είναι οι ποινικέ επιπτώσεις των ενεργειών μας. Διαπιστώνουμε ότι ορισμένοι πηγαίνουν από την Ευρώπη σε ζώνες συγκρούσεων ενδεχομένω ε, για να διαπράξουν τρομοκρατικέ ενέργειε όταν επανέλθουν στη χώρα του. Για παράδειγμα, η σφαγή στο Σαρλί Εμπντό. Πώ μπορεί ένα ε, εισαγγελέα να αποδείξει πέραν ε, αφιβολιών ότι κάποιος συμμετείχε σε εγκληματικές ε, ή πολεμικές ενέργειες σε μια ξένη χώρα και ότι έχει την πρόθεση να διαπράξει όταν θα επανέλθει στη χώρα του τρομοκρατικές ενέργειες. Πώς μπορούμε να το αποδείξουμε αυτό όταν δεν έχουμε ορισμό. Φυσικά είναι θέμα εξισορρόπησης μεταξύ των προσπαθειών για να μην έχουμε τρομοκρατικές ενέργειες στην Ευρώπη και του σεβασμού των ε, ε, δικαιωμάτων των ε, ατόμων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Είναι σαφές ότι πρέπει να δώσουμε μια ευρωπαϊκή απάντηση στην επίθεση της τρομοκρατίας και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο Συμβουλίου της Ευρώπης η καταπολέμηση αυτών των μαχητών ευρωπαϊκής προέλευσης θα είναι αποτελεσματική εφόσον υπάρξει κοινή αντιμετώπιση από πλευράς των κρατών μελών. Στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον προηγούμενο Φεβρουάριο ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ορίσει με σαφή τρόπο τους ε, μαχητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους Ευρωπαίους μαχητές, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την νομική επάρκεια της πρότασης. Η σύμβαση λοιπόν για την πρόληψη των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων θα είναι μια σωστή βάση εφαρμόζοντας και το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. ψήφισμα λοιπόν 2178 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ένα ψήφισμα το οποίο είναι απαραίτητο για να λάβουμε υπόψη μας και να μπορέσουμε να ασκήσουμε διώξεις σε νέες μορφές τρομοκρατίας όπως τα ταξίδια στο εξωτερικό για τρομοκρατικούς στόχους όπως και η χρηματοδότηση, στήριξη και διευκόλυνση τέτοιου είδους ε, αποστολών. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ε, συμπεριλάβουμε το πρωτόκολλο αυτό στο κοινοτικό δίκαιο, τότε θα έχουμε στη διάθεσή μας ένα ενιαίο κοινοτικό δίκαιο πέραν των, των συγκεκριμένων ε, συνεργασιών και να εναρμονίσουμε την απόκριση και αντίδραση της ποινική δικαιοσύνης απέναντι στους ξένους μαθητές. Συγγνώμη για την υψηλή ταχύτητα της παρέμβασής μου. Ο κ. Αγουιλάρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα στα πλαίσια της συζήτησης για τα πολιτικά θέματα και την έχουμε κάνει επανειλημμένα. Μόνο και μόνο τους τελευταίους μήνες. Δεν συζητάμε την τρομοκρατία σε πολιτικό επίπεδο, μιλάμε για την καταπολέμησή της σε νομικό επίπεδο. Και εδώ το θέμα είναι περίπλοκο και μάλιστα είναι το πιο περίπλοκο θέμα που έχω να αντιμετωπίσει εδώ και καιρό. Εγώ είμαι ε, νομικός, είμαι νομομαθής και νομοθέτης σε εισαγωγικά. Και νομίζω ότι αυτό το, αυτή η πρόταση η οποία γίνεται είναι η πλέον περίπλοκη που έχω συναντήσει. Υπάρχει ένα ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τους ξένους μαχητές. Μετά υπάρχει μια σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης όχι της Ευρωπαϊκής Ένωση, Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Μετά υπάρχει μια εντολή διαπραγμάτευση για ένα πρωτόκολλο, για μια απόφαση πλαίσιο, έτσι ώστε να τροποποιήσουμε την υπάρχουσα απόφαση πλαίσιο για την καταπολέμηση των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων. Έτσι ώστε να μπορέσουμε δηλαδή να προχωρήσουμε σε διώξει και να ποινικοποιήσουμε ενέργειες όπως η εκπαίδευση, η συμμετοχή σε εκπαίδευση, οι μετακινήσεις, τα ταξίδια ή η διάθεση, πρόθεση ε, μετακίνησης για τρομοκρατικούς στόχους. Το θέμα είναι θέμα νομικής ασφάλειας, όπως είπατε, ε, και μιλάω για τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με ποιο τρόπο το πρωτόκολλο αυτό θα μας δώσει τις παραμέτρους που απαιτούνται έτσι ώστε να υπάρξει νομική ασφάλεια απαραίτητη ε, για την αλλαγή των, ε, του ποινικού κώδικα σε κάθε χώρα μέλος, έτσι ώστε να υπάρξει ένα σαφές πλαίσιο αναφοράς που θα οδηγήσει στην πλήρη ποινικοποίηση τέτοιου είδους δραστηριοτήτων. Πέραν αυτού, υπήρξε μια ειδική συνάντηση του Συμβουλίου Υπουργών Νομικών Υποθέσεων αμέσως μετά τη σφαγή στο Παρίσι. Στη συνάντηση αυτή τα κράτη-μέλη πήραν την απόφαση να εκκινήσει μια νομοθετική πρωτοβουλία σε κάθε χώρα μέλος και σε κάθε κοινοβούλιο για την ποινικοποίηση τέτοιου είδους δραστηριοτήτων. Συνεπώς, σε επίπεδο νομικό, ποια θα είναι η προστιθέμενη αξία την οποία θα παράξει το συγκεκριμένο πρωτόκολλο, έτσι ώστε να επιτρέψει στις ισχύουσες διατάξεις να καλύψουν όλες ε, τις δραστηριότητες σε επίπεδο ποινικού δικαίου. Thank you, Chair. Ευχαριστώ για τη διαδικασία λήψη απόφαση. Δεν καταλαβαίνω πολύ καλά. Άκουσα τον κύριο Κουτσίκοφ και συνάγω ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης θα εγκρίνει τέλη Απριλίου την αναθεώρηση του πρωτοκόλλου και η υπογραφή θα γίνει 23 Μαΐου από τους Υπουργούς και κατά πάσα πιθανότητα και από τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Αλλά εδώ το Κοινοβούλιο πρέπει να παίξει το ρόλο του. Πρέπει να δώσει σύμφωνη γνώμη στα πορίσματα. Τι σύμφωνη γνώμη θα δώσουμε. Ενώ εντωμεταξύ διάφορα κράτη-μέλη θα έχουν ε, υπογράψει τις αλλαγές στη σύμβαση. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και νόμιζα επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τον ηγετικό ρόλο για τις διαπραγματεύσεις της Ένωσης με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Κάτι που θα μας επέτρεπε να εξετάσουμε την ε, εντολή της Επιτροπής πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Αλλά οι Υπουργοί Δικαιοσύνης και Εσωτερικών μας αφαίρεσαν αυτή τη δυνατότητα. Με προβληματίζουν όλα αυτά λοιπόν για τη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Και με προβληματίζει ο ρόλος μου. Πώς θα κάνω το δημοκρατικό μου καθήκον ως εκλεγμένος εκπρόσωπος να ελέγξω την εντολή και μετά να επικυρώσω. Ή όχι. Πραγματικά χρειάζομαι εξηγήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τη Λετωνική Προεδρία. Γιατί εγώ δεν νομίζω ότι είναι σωστή η αλληλουχία των ενεργειών. Βεβαιασμένα οδεύουμε προς ένα νέο πρωτόκολλο που μπορεί να είναι πολύ σημαντικό. Που μπορεί να έχει ως συνέπεια να παραβιαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα ορισμένων. Οπότε να επαναλάβω τις ερωτήσεις της ε, Σοφίνετφελντ. Νετφέλντ. Πώς θα αποδείξουμε την πρόθεση κάποιου. Ότι προτίθεται να πάει να εκπαιδευτεί για να διαπράξει τρομοκρατικές ενεργές. Θυμάμαι ότι κάποιοι Ολλανδοί πολίτες ταξίδευαν με ένα αυτοκίνητο στη Γερμανία και στο Port Bagage είχαν στρατιωτικές ε, στολές. Πώς είναι δυνατόν να συλλάβουμε κάποιον επειδή έχει στο πόρτ του ένα, μια στρατιωτική στολή, γιατί ίσως πήγαινε στη Συρία. Και αυτό αποφάσισε και ο Ολλανδός δικαστής. Δεν μπορείς να τους καταδικάσεις για προπαρασκευή τρομοκρατικών πράξεων. Και κάτι ακόμη. Ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών. Για να είμαστε σε θέση να συλλάβουμε έναν ύποπτο τρομοκρατικό ενεργειών. Καταλαβαίνω την ανάγκη γι' αυτό. Αλλά πώς θα διασφαλίσουμε ότι δεν ανταλλάσσουμε πληροφορίες από ένα ευρωπαϊκό κράτη, κράτος μέλος σε ένα καθεστώς που αντιλαμβάνεται πολύ διαφορετικά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πώς θα διασφαλίσουμε ότι αυτό το καθεστώς δεν θα ζητήσει να του παράσχουμε στοιχεία που δεν πρέπει να του δώσουμε ή τα οποία θα χρησιμοποιήσει με λάθος τρόπο. Ευχαριστώ, Ιούντιτ. Η κυρία Γκόμερ. Χθες ακούσαμε εδώ πέρα τον ε, επικεφαλής του Φράντεξ, ο οποίος παραδέχτηκε ότι τα κράτη-μέλη δεν κάνουν τίποτα. για να συλλαμβάνουν διακινητές ε, προσώπων. Και ξέρουμε ότι η εμπορία προσώπων, η διακίνηση προσώπων ε, είναι ποινικοποιημένη στο διεθνές δίκαιο, σε εθνικό δίκαιο, περιφερειακό δίκαιο και συνδέεται μάλιστα με την τρομοκρατία όλο και περισσότερο. Και τώρα προτείνουμε να ποινικοποιήσουμε πράγματα που σε πολλά κράτη είναι ήδη ποινικά αδικήματα γιατί η τρομοκρατία φυσικά είναι ποινικό αδίκημα. Η προστιθέμενη αξία αυτού του αναθεωρημένου πρωτοκόλου υποθέτω δεν είναι μόνο η εναρμόνιση και η κωδικοποίηση αυτής της ποινικοποίηση, αλλά και ταχύτερη έκδοση για τις χώρες που συμμετέχουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Αλλά έχει το αρνητικό που είπε μόλις η κυρία Σαρχεντίνη κάποια μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης θα μπορούσαν να κάνουν κατάχρηση αυτών των ενιών και των δυνατοτήτων που εισάγουμε. Α, βλέπουμε ότι το ένταλμα σύλληψη πολλέ φορέ χρησιμοποιείται με λάθο τρόπο για να συλλαμβάνονται διάφοροι αγωνιστέ υπέρ τη στήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν θα βοηθούσε ορισμένες κυβερνήσεις χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης που χρησιμοποιούν με λάθος τρόπο. Και τι προσταθεμένη αξία έχει για μας. Πώς θα συμβάλλει στο πιο σημαντικό, που είναι κατά τη γνώμη μου, η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών μας και εντός της Ένωσης και με τρίτες χώρες. Δεν βλέπω να έχετε εργαστεί αρκετά προς αυτή την κατεύθυνση που αυτό θα ήταν το πιο ουσιώδε στοιχείο. Σας παρακαλώ λοιπόν. Εξηγήστε μας. Σε τι βαθμό θα ενισχύσετε την ανταλλαγή προφοριών αλλά με σκόπιμο τρόπο που να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως τα αντιλαμβανόμεθα. Αναφερθήκατε τη CIA και το ρόλο του Κοινοβουλίου. Αλλά και μέχρι σήμερα οι κυβερνήσει μα δεν έχουν αποδεχτεί την ευθύνη του για το θέμα αυτό. Στη χώρα μου, για παράδειγμα, την Πορτογαλία, οι μυστικέ υπηρεσίε δεν έχουν δικαίωμα καθόλου να ακούνε ε, ηλεκτρονικές συνομιλίες αλλά το κάνουν το είδαμε σε μια σε μια υπόθεση πρόσφατα σε ένα δικαστήριο υπάρχουν πολλές αντιφάσεις Δεν καταλαβαίνω σε τι βαθμό και με τι τρόπο αυτό θα μας βοηθήσει στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η κυρία Μάια. Χολμάια. Μάια, συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ρωτήσω κάτι για το άρθρο 4 του πρωτοκόλου που αναφέρεται στα ταξίδια στο εξωτερικό. Και αναρωτιέμαι, Ίσως θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε περισσότερο τι γίνεται με την περίπτωση ανθρώπων που έχουν διπλή υπηκότητα και πηγαίνουν σε μια χώρα της οποίας επίσης έχουν την υπηκότητα. Αυτό συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο αυτό ή όχι, αυτή η περίπτωση. Τώρα, κυρία Χολμάιερ. Ω συντονίστρια του ΕΛΚ δεν θέλω μόνο να επικρίνω για κάτι διαφορετικό, λοιπόν, με διαφορετικό τρόπο θα μιλήσω. Θέλω να ευχαριστήσω το Συμβούλιο της Ευρώπης για, τον, ε, για την πόση δουλειά έκανε για να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα. Βεβαίως ε, έχω κάπως ε, κριτική άποψη, αλλά έναντι των κριτικών των συναδέλφων Ιντφελτ και Σαργεντίνη. Δεν μπορούμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τη μία μεριά να επικρίνουμε τα κράτη-μέλη ότι αφήνουν ορισμένους να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για να κάνουν σοβαρά εγκλήματα και μετά όταν σκεφτόμαστε Πώς είναι δυνατόν να ε, διαπιστώσουμε την ταυτότητα κάποιου που μπορεί να έχει αυτή την πρόθεση και να το σταματήσουμε, να επικρίνουμε και αυτός προσπαθούν να το κάνουν αυτό. Εγώ θα ήθελα να δω υπό ποιε προϋποθέσεις θα ήταν δυνατόν τα κράτη-μέλη να καθορίσουν κάποιους κανόνες για το τι σημαίνει κάποιος που προσπαθεί να πάει κάπου, πώς θα δημιουργήσουμε κανόνες για το πώς θα διαπιστώσουμε την ταυτότητά του, ούτως ώστε να σταματήσουμε αυτούς που θέλουν να κάνουν ταξίδια για να διαπράξουν σοβαρά εγκλήματα. Και δεύτερον, το, το θέμα της σχέσης ε, του Ισλαμικού κράτους και του οργανωμένου εγκλήματος, η Σνάλφος Γκόμες μίλησε για την εμπορία τόμων, υπάρχουν πολλοί στενές διασυνδέσεις και ξέρετε ότι στη Λιβύη το Ισλαμικό κράτος έχει στην ουσία τα λιμάνια ε, στα χέρια του. Τι προτείνει το Συμβούλιο της Ευρώπης για να ληφθεί και αυτό υπόψη. Πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε αυτές τις ε, διασυνδέσεις μεταξύ της διεθνούς τρομοκρατίας και του οργανωμένου κλίματος. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Φαγιώνη Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω τα σχόλια και τις ερωτήσεις τις οποίες έκαναν οι προηγούμενοι συνάδελφοι. Να αναφερθώ σε ένα άλλο θέμα όμως. Το θέμα αυτών οι οποίοι επανέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Των πολιτών που επιστρέφουν. Θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τους επιστρέφοντες στις χώρες μας. Έχουμε το μέτρο της κατάσχεσης των διαβατηρίων Έχουμε ακόμα και το μέτρο της αφαίρεσης της ευρωπαϊκής υπηκότητας, αλλά αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Πρέπει να γίνει μια συζήτηση για να δούμε με ποιο τρόπο θα τα συζητήσουμε αυτά, θα, θα προχωρήσουμε στον τομέα αυτό, τι μέτρα θα πάρουμε. Και θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε με αποτελεσματικότερο τρόπο την προπαγάνδα των τρομοκρατών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο θα ήθελα πιο συγκεκριμένες προτάσεις you. Uh, Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ το Συμβούλιο για τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε. Ιδιαίτερα το θέμα πώς μπορούμε να, να αναλάβουμε προληπτικές ενέργειες. Δεν βλέπω στο κείμενο να έχετε σκεφτεί τα προληπτικά μέτρα πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ριζοσπαστικοποίηση Δηλαδή να εμποδίσουμε να σκεφτούν να γίνουν μαχητές. Βεβαίως πρέπει να το κάνουμε και μέσω παρέμβασης στο διαδίκτυο. Και ακούσαμε για την ανταλλαγή προφοριών. Βεβαίως. Βεβαίως. Υπάρχει αυτή η ανταλλαγή γενικά πληροφοριών, αλλά θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τους ξένους μαχητές, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα κινητικοί και με πολύ έξυπνο τρόπο και με διάφορα τεχνάσματα κάνουν τις μετακινήσεις τους. Πρέπει να δούμε πώς θα συνεργάζονται και τι στοιχεία θα ανταλλάσσουν οι υπηρεσίες. Είναι τα στοιχεία για τα ταξίδια, τα τραπεζικά στοιχεία και οι διάφορες επικοινωνίες. Εδώ λοιπόν πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι για να ανακαλύψουμε ποιοι έχουν την πρόθεση να γίνουν ξένοι μαχητές και ποιοι προσπαθούν να τους ριζοσπαστικοποιήσουν. Πρόεδρος. Ωραία. Έδωσα το λόγο σε όλους τους ε, συναδέλφους. Να επανέλθω προς τους ε, εμπειρογνώμονές μας ε, με την ίδια σειρά. Πρώτος ο κύριος Λόικ. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να τα κατηγοριοποιήσω. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Πρώτον, για την πρόθεση. Πολύ σημαντικό στοιχείο. Και μας έχει απασχολήσει ιδιαίτερα. Το αναφέρατε ορισμένοι. Η Ευρωπαϊκή Ποινική Νομοθεσία και το Εθνικό Νομικό Σύστημα δεν διώκει προθέσεις αλλά μόνο ενέργειες. Ωστόσο, ωστόσο για την τρομοκρατία ακόμη και η απόφαση πλαίσιο η δική μας κάνουμε μια διάκριση. Πρέπει να κάνουμε διαχωρισμό μεταξύ της νομότυπης χρήσης ορισμένων διαδικασιών και της παράνομης. Γι' αυτό έχουμε κάποια στοιχεία που λένε ότι μπορεί να είναι η προετοιμασία μιας πράξης, χρηματοδότηση, κατάρτιση μια πράξη με την πρόθεση να σκοτώσετε, να τρομοκρατήσετε τον πληθυσμό, να επηρεάσετε παράνομα τις δημόσιες πολιτικές, τις πολιτικές των κυβερνήσεων. Αυτά λέει η απόφασή μας στον τομέα της τρομοκρατίας λοιπόν. Πρέπει να έχουμε αντικειμενικά στοιχεία βέβαια, μια ενέργεια, μια συμπεριφορά μαζί με την πρόθεση. Γιατί ακοντράριο αυτό που δεν θέλουμε είναι ότι ένας που νομότυπα χρησιμοποιεί ένα όπλο ή εκρηκτικά και τα μεταφέρει γιατί για παράδειγμα εργάζεται στην εξόριξη ή αυτοί που ταξιδεύουν νομότυπα τέθηκε το θέμα της διπλής υπηκότητας αν πάω λοιπόν πίσω στη χώρα προέλευσης της μητέρας μου ή στη χώρα του δεύτερου διαβατηρίου μου αυτό είναι νομότυπη μετακίνηση δεν θα υπάρχει τίποτα παρά, παράνομο. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικά στον ορισμό της τρομοκρατία, που τον έχουμε ήδη στην απόφαση πλαίσιο, να έχουμε αυτά τα δύο στοιχεία. Πρέπει να υπάρχει και αντικειμενική ενέργεια και συμπεριφορά, αλλά μπορεί να μην αρκεί. Γιατί αλλιώ θα ήταν ε, ε, πολύ ευρεία η και θα διώκαμε και άτομα τα οποία συμπεριφέρονται ή προβαίνουν σε κάποιες ενέργειες ε, νομότυπα. Για παράδειγμα, στην εξορυκτική, στον εξορυκτικό κλάδο, οι ένοπλες δυνάμεις. Νομότυπα χρησιμοποιούν όπλα, κάποιες τεχνικές. Αυτή είναι η γραμμή. για παραδειγμα στην στον είναι λεπτή, αλλά πρέπει να χαραχθεί. Και μετά βέβαια το θέμα θα είναι, στα πλαίσια των εθνικών ποινικών διαδικασιών, θα τίθεται το θέμα τι αποδεικτικά στοιχεία έχουμε. και όλες οι ανακριτικές και ιδιοκτικές τεχνικές με βάση τις ε, συνταγματικές μας παραδόσεις και τα θεμελιώδη δικαιώματα σε κάθε χώρα θα πρέπει να αξιοποιούνται και δεν αλλάζει τίποτα. Δεύτερον, κύριε Λόπεθ Αγγιλάρ, είναι πολύ περίπλοκη η κατάσταση. Είναι σαν λαζάνια σε στρώσεις. Ωραία, ωραία. Ακούγεται ένας ύμνος όταν μιλάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λοιπόν, τι έλεγα. Και δεν είναι ευθύνη του κυρίου Κούτσικοφ. Ε, είναι μια πολύ περίπλοκη κατάσταση που δεν δημιουργήσαμε εμείς, αλλά την οποία πρέπει να χειριστούμε. Και έχει επιπτώσεις και στη χρονική αλληλουγία. Είχαμε την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Μετά το Συμβούλιο της Ευρώπης αντέδρασε πολύ γρήγορα στις 21 Ιανουαρίου ξεκίνησε αυτή τη νέα εργασία ενώ ήδη συζητούσαμε όπως ξέρετε στο Συμβούλιο με λεπτομέρειες πώς πρέπει να αναθεωρήσουμε τα κείμενά μας για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο των ξένων μαχητών σε ενωσιακό πλαίσιο. Και αυτά τα δύο συνέπεσαν λόγω της πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης και η τέταρτη στρώση τα λαζάνια στα λαζάνια είναι κάποια κράτη-μέλη που ανέλαβαν νομοθετικές πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο. Είναι δύσκολη κατάσταση λοιπόν. Ο χρόνος πιέζει ιδιαίτερα και πρέπει όλα αυτά να ενταχθούν σε ένα ενιαίο και συνεπές πλαίσιο. Τώρα τι θα γίνει μετά και πώς αυτό θα επιδράσει στον ενωσιακό και εθνικό νόμο, αυτό θα το δούμε. Γι' αυτό είπα ότι στην εντολή μας υπάρχει μία ρήτρα αποσύνδεσης. Δηλαδή για την Ένωση και τα κράτη-μέλη λέμε θα κάνουμε μεταξύ μας ό,τι μπορούμε αξιοποιώντας τον ενωσιακό και εθνικό νόμο. Αυτό ίσχυε και με βάση το άρθρο 26 της αρχικής σύμβασης, το οποίο ακριβώς αντιγράψαμε στην εντολή μας και στο πρωτόκολλο για να έχουμε κάποιο περιθώριο να συζητήσουμε μεταξύ μας εάν θα τροποποιήσουμε για παράδειγμα την απόφαση πλαίσιο ή θα αφήσουμε τα κράτη-μέλη εθνικά να το ρυθμίσουν. Αυτή η συζήτηση θα γίνει μετά γενέστερα. Τώρα, οι προθεσμίες, η υπογραφή, η κατάληξη. Κατανοώ λέτε κυρία μου. Γιατί ξέρετε η ζωή μας ήταν μια κόλαση μαζί με την Προεδρία από νομική άποψη ξέρετε είναι πολύ απαιτητικά αυτά τα θέματα γιατί μερικές από τις έννοιες που συζητήσαμε για την ποινικοποίηση κάποιων συμπεριφορών υπάρχουν ήδη ε, διατάξεις που έχουμε γκρίνει για αυτό από το 2008 και μετά αλλά είναι η πρώτη φορά που στην περίοδο μετά τη Λισαβόνα, μετά την πενταετή δηλαδή μεταβατική περίοδο, είναι η πρώτη φορά που ε, οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται και εξωτερικά. Στα πλαίσια δηλαδή του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είμαστε λοιπόν πεπισμένοι με βάση αυτά που προανέφερα ότι με βάση τη νέα συνθήκη της Λισαβόνας όλα αυτά είναι αποκλειστική ενωσιακή αρμοδιότητα. Αλλά κάποια κράτη-μέλη δεν συμμερίζονται αυτή την άποψη. Οπότε ένα τμήμα του πρωτόκολλου μπορεί να είναι σε ε, κοινή αρμοδιότητα. Αυτό για το ότι πρέπει να είμαστε συνεχώ σε επαφή. 24 ώρε 7 μέρε την εβδομάδα. Α το αφήσουμε λοιπόν ε, κατά μέρο αυτό. Α δράσουμε από κοινού στο Στρασβούργο, η Κομισιόν να συντονίζει τη διαπραγμάτευση, να συμμετέχουν τα κράτη-μέλη και στην πράξη στι τρει συναντήσει για διαπραγματεύσει που ανέφερε ο κ. Κούτζικοφ λειτουργήσε πολύ καλά. επίση αποφασίσαμε ότι κατόπιν θα κάνουμε μια πιο τεκμηριωμένη και πολύ πιο γαλήνια συζήτηση για να προσπαθήσουμε να διαχωρίσουμε τι είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης και τι είναι κοινή αρμοδιότητα. Αυτή η συζήτηση θα γίνει όταν θα έχουμε το σχέδιο απόφαση του Συμβουλίου για την κατάληξη και υπογραφή του πρωτοκόλλου. Έτσι δίνουμε λίγο χρόνο στον εαυτό μας για να κάνουμε μια πιο λιγότερο βεβιασμένη συζήτηση με πλήρη γνώση των στοιχείων και με τον έλεγχο του Κοινοβουλίου για την ανταλλαγή προφοριών θα σας εξηγήσω ο κύριος Κουτζίκοφ αλλά μόνο το εξή. πρόκειται απλώ και μόνο να δημιουργήσουν οι χώρες μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης τα αναγκαία σημεία επικοινωνίας για να μπορούμε ανα πάσα στιγμή να ανταλλάξουν πληροφορίες όταν κάποιος διαπιστώνεται ότι επιδιώκει να διασχίσει κάποια σύνορα για να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο των ξένων μαχητών. Εκπεφρασμένα λέμε, και αυτή ήταν η διαπραγματευτική μας άποψη, ότι αυτό δεν προκαλεί νέες υποχρεώσεις ανταλλαγής στοιχείων. Είναι απλώς η δημιουργία σημείων επαφής δεν αποδεχόμεθα καμία νέα υποχρέωση ανταλλαγής προσωπικών δεδομένων. Τι θα γίνει στην Ευρώπη. Δεν θα γίνει τίποτα. Για τα κράτη-μέλη ήδη έχουν αυτά τα σημεία συνεχούς επαφής. Τώρα για τους επιστρέφοντες και τα ευρύτερα θέματα. Τους επιστρέφοντες πολίτες της Ένωσης και τη δικτύωση, τη διασύνδεση. Το λέει το άρθρο 6 του πρωτοκόλλου όπου αναφερόμεθα σε όλα αυτά τα δίκτυα και τους ε, αυτούς που κάνουν ε, που διευκολύνουν που δεν καταρτίζουν ε, μαχητές δεν διαπράττουν ενέργειες αλλά βοηθάνε άλλους να τα κάνουν αυτά τα λέει το άρθρο 6 για το ευρύτερο θέμα που θέσατε τι θα κάνουμε με τους επιστρέφοντες Έχουμε σκεφτεί τίποτα για εναλλακτικέ λύσεις προς την ε, φυλάκιση. Ναι, υπάρχουν τέτοιες ε, συζητήσεις. Στη συζήτηση που, κάνουν, ε, που κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τίθεται το ερώτημα. Όλοι αυτοί οι έχει έννοια να φυλακίζονται. Ορισμένοι που επιστρέφουν είναι πράγματι εγκληματίες και διεκδικούν τις πράξεις τους. Αλλά πολλοί έχουν απλώς αειδιάσει ε, υποφέρουν από μετατραυματικό σύνδρομο. Σκεφτόμαστε λοιπόν με το Συμβούλιο Υπουργών, με τη Σύμβαση για την Καταπολέμηση της Δημοκρατίας. Είναι ευρύτερο αυτό το θέμα, προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε. Και για το ίντερνετ βέβαια είναι πολύ δύσκολο αυτό το θέμα. Δεν προτιθέμεθα και δεν πιστεύουμε ότι η ρυθμιστική άποψη σε νοσιακό επίπεδο θα ήταν η καλύτερη, θα ήταν η κατάλληλη, αλλά το να ε, εντοπίσουμε το παράνομο περιεχόμενο στο ίντερνετ και επίσης να απαντάμε σε κάποιες ε, ε, ιστοσελίδες προπαγάνδας Έχουμε αρχίσει την ενέργεια, τις ενέργειες μας γι' αυτό, έχουμε κάνει δύο συναντήσεις, θέλουμε να κάνουμε ένα διαθρωμένο διάλογο σε πιο λειτουργικό επίπεδο. Έχουν γίνει λοιπόν δύο συζητήσεις και με την κυρία Μέλστρομ, πώς να αξιοποιήσουμε τις κοινότητες χρηστών, μαζί δηλαδή με τους ε, χρήστες του ίντερνετ, να αξιοποιήσουμε και τις δικές τους δυνατότητες να αναφέρουν τέτοιο περιεχόμενο. Και αυτή η ιδέα να υπάρχει μία μονάδα για να ε, ψάχνει το περιεχόμενο του ίντερνετ, ούτως ώστε το παράνομο, το παράνομο περιεχόμενο να εντοπίζεται και μετά να δούμε τι θα γίνει με αυτό το περιεχόμενο. Να το στέλνουμε πίσω στους παρόχους, για παράδειγμα, να το, να το εντοπίσουμε στους παρόχους για απόσυρση. Μια τεχνική ερώτηση. Αυτό σημαίνει ότι το πλαίσιο του 2008, της ασφάλειας του 2008 χρειάζεται να αναθεωρηθεί ή όχι. Είναι μια δυνατότητα. Είτε θα το κάνουμε αυτό με μια οδηγία μετά τη συνθήκη ή θα το κάνουμε σε εθνικό επίπεδο. Thank you very much. Um, είναι πολύ δύσκολο να προσθέσει κανείς κάτι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλυψε το σύνολο περίπου των ερωτήσεων από τα κράτη-μέλη. Τώρα, το Συμβούλιο και η Προεδρία θέλουμε να υπογραμμίσουμε μόνο ότι το πρωτόκολλο τη σύμβαση αυτή είναι κάτι το οποίο δέχονται τα κράτη-μέλη. Θεωρούν τα κράτη-μέλη, εκτιμούν ότι είναι μια καλή βάση για μια ελάχιστο ε, επίπεδο εναρμόνιση. Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ένα διαφορετικό όργανο βέβαια, ένας διαφορετικός θεσμός, έχει 80 τόσα μέλη. Έχει 56 μέλη και έτσι κάθε ένα από τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης εφόσον το επιθυμεί μπορεί να αποδεχθεί το συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Η προστιθέμενη αξία του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου λοιπόν είναι ότι καλύπτει όχι μόνο τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά εφόσον το επιθυμούν και χώρες εκτός αυτής. Αυτό διασφαλίζει η σωστή λειτουργία του συστήματος των εκδόσεων αλλά και της αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής. Είναι κάτι το οποίο συνδέεται και με την αρχική σύμβαση, τη μητρική λεγόμενη σύμβαση, αλλά και με τα προηγούμενα πρωτόκολλα. Αν κάποιες χώρες δεν θέλουν να συνδεθούν, το μόνο που, θέλουν, που πρέπει να κάνουν είναι να μην αλλάξουν τις ισχύουσες ρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο. Οι χώρες μέλη λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχουν σε διαδικασίες του Συμβουλίου της Ευρώπης θα πρέπει και εμείς ε, ε, σε σχέση με την θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Συμβούλιο της Ευρώπης να αναλάβουμε το ρόλο που μας αναλογεί. Το θέμα είναι να προσπαθήσουμε να δούμε τι είδους αρμοδιότητα υπάρχει εδώ, αν υπάρχει αποκλειστική αρμοδιότητα ή αν υπάρχει διαμερασμένη αρμοδιότητα ανάμεσα στα κράτη-μέλη ε, και την Ευρωπαϊκή Ένωση, την κοινότητα και το πώς αυτό εκφράζεται στο εσωτερικό του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η προηγούμενη οδηγία θυμίζω ότι δεν καλύπτει τις μετακινήσεις, τα ταξίδια, γιατί είναι ένα φαινόμενο νέο σχετικά. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να δούμε ποια είναι τα τμήματα της πρότασης αυτής τα οποία θα ανήκουν στο καινούριο συμπληρωματικό πρωτόκολλο και ποια θα είναι αυτά τα οποία δυνητικά μπορεί να ολοκληρωθούν και να πάρουν συγκεκριμένη μορφή σε εθνικό αποκλειστικά επίπεδο. Αυτή είναι η πορεία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ε, για να καταλήξουμε στο νέο πρωτόκολλο. Το Συμβούλιο της Ευρώπης λοιπόν παίζει τώρα πλέον ένα πολύ σημαντικό ρόλο και προσθέτει αξία και στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα για την πιθανότητα μιας νέας οδηγίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα αξιολογήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κρίνει ε, σε επίπεδο Συμβουλίου Υπουργών τι θέσεις έχουν εκφράσει τα κρατη Δεν έχει υπάρξει ομοφωνία πλήρως και δεν γνωρίζουμε αν θα χρειαστούμε ένα νέο ε, κοινοτικό νομικό μέσο. Εφόσον τα κράτη-μέλη επιθυμούν, είναι σε θέση απλά να προσυπογράψουν το συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Εγώ δεν ξέρω πότε θα ανοίξει η διαδικασία των υπογραφών. Τουλάχιστον δεν είμαι ενήμερη γι' αυτό. Αλλά πάντως οι διαδικασίες είναι γνωστές που θα ακολουθηθούν από εδώ και πέρα όπως επίσης είναι σαφής και ο ρόλος τον οποίο μπορεί να παίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υπογραφή. Μέχρι τώρα μιλούσαμε για την εντολή για τη διαπραγμάτευση. Δεν μιλήσαμε για τη διαδικασία εντολής για την υπογραφή του πρωτοκόλου. Είναι ένα θέμα το οποίο θα απαιτήσει χρόνο για συζήτηση στο Συμβούλιο. Λοιπόν, προς το παρόν δεν αλλάζει κάτι. Τουλάχιστον έτσι κρίνει η Προεδρία του Συμβουλίου. Βλέπω ότι και οι δύο ζητάτε το λόγο. Αλλά να σας πω ότι θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Κοιτάξτε, για διαδικαστικό ζητάω το λόγο, λέει η κυρία Σαρτζεντίνη. Κοιτάξτε, δεν μιλάω για την ουσία, μιλάω για τη διαδικασία. Εμείς ζητάμε κάποιες διευκρινήσεις για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Δεν έχει διευκρινιστεί η διαδικασία ανάμεσα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, ποιο έχει αποκλειστική αρμοδιότητα και για ποιο τομέα. Όσο δεν διευκρινίζεται αυτό, τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να υπογράψουν. Δεν μπορούν να υπογράψουν αν δεν ολοκληρώσουμε και εμείς σαν κοινοβούλιο ε, το τι ε, πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, το θέμα συζητιέται στους διαδρόμους, αλλά δυστυχώς εγώ σαν βουλευτής δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου. Κυρία Ιντβέλτ. Θα ήθελα η Γραμματεία να μας δώσει ένα σημείωμα το οποίο να υπογραμμίζει ακριβώς το ποια είναι η διαδικασία, ποιες είναι οι προθεσμίες, ποια είναι η κατανομή των αρμοδιοτήτων. Όλα αυτά πρέπει να διευκρινιστούν. Κοιτάξτε, η διαδικασία που ακολουθείτε είναι η πιο συγκεχημένη και μπερδεμένη που έχω δει εγώ ποτέ μου στο Κοινοβούλιο. Και μιλάμε για ποινικοποίηση συμπεριφορών και για πιθανή ποινικοποίηση μια απλή αντικειμενικής πράξης μετακίνησης ενός ταξιδιού. Μιλάμε δηλαδή για κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σοβαρό. Περιμένω λοιπόν διευκρινήσεις από τη γραμματεία το ταχύτερο δυνατόν να διευκρινίζει η γραμματεία σε ποια φάση βρισκόμαστε και ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε. Η Επιτροπή έχει το λόγο. Δεν διαφωνώ, δεν γυρνάω γύρω-γύρω από το θέμα, είμαι σαφής πιστεύω. Χρειαζόμαστε επιγόντως την εντολή αυτή. Αν δεν την έχουμε, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα συμφέροντά της δεν θα συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις αυτός είναι ο στόχος τακτικής. Είμαστε πρακτικοί, είμαστε ενωμένοι, οι συνάδελφοι και ο κ. Κούτικοφ το επιβεβαιώνει αυτό. Με την Προεδρία έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ καλά έτσι ώστε ενωμένοι να προχωρήσουμε. Πράγματι όμως, εξαιτία του χρονικού πλησίου, Αλλά και πάλι δεν είναι κάτι που δημιουργήσαμε εμείς. Συμβαίνει. Το Συμβούλιο της Ευρώπης ανέλαβε την πρωτοβουλία και εμείς θέλουμε να συμμετέχουμε. Δεν μπορούμε να σιωπούμε, να είμαστε ανύπαρκτοι. Σίγουρα υπάρχουν περιορισμοί και ζητώ συγγνώμη. Είναι όμως μια κατάσταση που προσπαθούμε να διορθώσουμε. Εμείς, η Επιτροπή, η Προεδρία δεν δημιουργήσαμε αυτή την κατάσταση. Πράγματι, είναι γραπτά στην εντολή ότι όλοι συμφωνούν. Υπάρχουν θέματα που είναι κοινοτική αρμοδιότητα. Υπάρχουν θέματα, και εδώ αναφέρομαι στα σημεια επαφη επαφής 24-7, που είναι η επιμερισμένη ή η εθνική αρμοδιότητα. Τι θα κάνουμε όμως, θα το αυτό τώρα όταν ο χρόνος περνάει και την επόμενη εβδομάδα είμαστε στο επόμενο στάδιο. Όχι, γραπτά στην εντολή λέμε ότι αυτά τα θέματα τα αφήνουμε και θα επανέλθουμε όταν έχουμε το σχέδιο του Συμβουλίου προς υπογραφή. Αυτό που ζητάτε κι εσείς. Συζητήσεις λοιπόν θα γίνουν πριν υπογράψει οποιοδήποτε. Θα γίνει η συζήτηση αυτή. Ελπίζω αυτό να σας βοηθάει. σε ευχαριστούμε. Ο κύριος Κοτσικόφ τώρα και παρακαλώ προσπαθήστε να είσαστε σύντομος, όσο γίνεται πιο σύντομος. Ευχαριστώ πολύ. Τηλεγραφικά λοιπόν. Δεν θα ασχοληθώ με τα θεσμικά ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μόνο που μπορώ να πω ότι η ομοιρία για παράδειγμα είναι έγκλημα. Μην με βάρετε όμοιρο λοιπόν για θεσμικά ζητήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους ευρωβουλευτές για όλα τα σημεία που έθιξαν, ιδιαίτερα αξιόλογα, όλα. Μερικά δεν έχουν να κάνουν όμως με το πρωτόκολλο. Ο λόγος για τον οποίο το πρωτόκολλο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει γρήγορα είναι γιατί έχει ένα περιορισμένο εύρο εφαρμογή. Δεν ασχολείται με θέματα παρακολούθησης, με θέματα πρόληψης, με θέματα ριζοσπαστικοποίηση. Δεν έχω χρόνο να σα πω τι κάνει για αυτά το Συμβούλιο της Ευρώπης, αλλά δεν πρόκειται για αυτά. Να επικεντρωθούμε στο πρωτόκολλο παρακαλώ, όσον αφορά την ποινικοποίηση τη πρόθεση. Δεν υπάρχει ποινικοποίηση της πρόθεσης. Τελεία και παύλα. Ούτε στην αρχική σύμβαση ούτε στο πρωτόκολλο. Τελεία. Στο ποινικό δίκαιο. Στην Ευρώπη για τα περισσότερα αδικήματα υπάρχει η πρόθεση και η πράξη. Πολύ λίγα αδικήματα, μάλλον πολύ λίγες πράξεις γίνονται χωρίς πρόθεση. Αλλά δεν υπάρχει ποινικοποίηση της πρόθεσης αυτής καθευτής. Δεν υπάρχει στο ποινικό δίκαιο αυτό ούτε στις χώρες μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το πρωτόκολλο λοιπόν δεν ποινικοποιεί την πρόθεση. Δεν έχω χρόνο τώρα να επεκταθώ περισσότερο. Εξηγούνται όμως όλα πιστεύω στο επεξηγηματικό σκέλος. Ένα από τα ζητήματα τα οποία δημιουργεί πρόβλημα, αλλά δεν το λύνει έτσι καλώς το πρωτόκολλο, είναι το θέμα των ορισμών. Τι είναι τρομοκρατία. Αυτό αναφέρεται αλλού. Τέλος, και πάντα πολύ τηλεγραφικά για τα σημεία επαφής 24-7, ή μάλλον πριν φτάσω στο 24-7. Το να ταξιδεύει κανείς με στόχο ή μάλλον το πρωτόκολλο δεν κοιτάει μόνο αυτούς οι οποίοι θα επιστρέψουν, αλλά αυτούς που θα ταξιδέψουν για να πάνε να ενταχθούν σε μια τρομοκρατική οργάνωση. Και τώρα έχουμε στο 24 λεπτά. Πρόκειται για ανταλλαγή πληροφοριών στην αστυνομία. Δεν πρόκειται για συνθήκη έκδοσης, δεν πρόκειται για την αμοιβαία συνδρομή, τίποτα τέτοιο. Πρόκειται απλώς και μόνο πολύ περιορισμένα πληροφορίες της αστυνομίας που θα μπορεί να ενημερώνει στα σύνορα για να μπορούν να κρίνουν οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί επί τόπου. Το πρωτόκολλο αυτό έχει σαν στόχο να αντιμετωπίσει ένα ζήτημα επίκαιρο και που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν προσπαθεί και δεν είναι δυνατόν να λύσει όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την τρομοκρατία που υπάρχουν και δυστυχώ φοβάμαι θα συνεχίσουν να υπάρχουν για κάποιο διάστημα τουλάχιστον. Πρόεδρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η γραμματεία ε, ζητήθηκε να ετοιμάσει ένα σημείωμα. Θα επανέλθουμε σε αυτό λοιπόν όταν θα έχουμε νέες εξελίξεις και όταν θα ζητηθεί, θα έρθει σε μας, δηλαδή το αίτημα για σύμφωνη γνώμη. Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Ευχαριστούμε που ήρθατε στη συνεδρίασή μας και για την ε, συνεργασία σας αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε τη συνεδρίασή μας από κοινού με την Επιτροπή ΔΕΒΕ στην αίθουσα 3G3 στο κτίριο Αλτιέρο Σπιρέλη. Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας θα λάβει χώρα στις 13 Απριλίου, 3 με 6.30 το απόγευμα και 14 Απριλίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12.30 και μετά 3 με 6.30. Ευχαριστώ πολύ. Για όσους δεν έρθετε στην κοινή συνεδρίαση, σας εύχομαι καλό Πάσχα.